της Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι κάνει τώρα. Εκατοντάδες χιλιάδες ε, του σε άσυλο είναι ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νόμιμοι πλέον, επομένως ε, πρέπει να δείξουμε και αλληλεγγύη προς αυτούς, μέτρα υγείας και για αυτούς. Αλλά διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στέλνει ε, χρήματα για άλλες πανδημίες, για παράδειγμα σε επιδημίες ελονοσίας. Ε, ε, αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει δισεκατομμύρια ευρώ σε αναπτυσσόμενες χώρες για τον κορονοϊό. Ξέρετε, σε αυτό το απίθμενο πηγάδι την Αφρική, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία έχουν τεράστια προβλήματα για τον κορονοϊό, αλλά απλώς τους δίνουν ψίχουλα. Η Φλάνδρα μόλις πήρε 6 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει τι σημαίνει ευρωκράτος, ευρωπαϊκή γραφειοκρατία αναφέρονται σε ανθρωπιστικά μέτρα για όλο τον κόσμο, αλλά κάθε φορά που απειλείται η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυγχάνει. Καλύτερα προτιμούν να κάνουν πράγματα για κόσμο εκτός... Ε, Ευχαριστούμε κύριε Ντεμάν. Ακολουθεί για ένα μισή λεπτό ο κύριος Φανόβερθελτ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, ε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής ε, και να πω δύο λόγια για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, τις οικογένειές τους ε, και όλους αυτούς που εργάζονται στα συστήματα υγείας και τις προσπάθειες αυτών των ανθρώπων ε, για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θα οδηγήσει φυσικά σε μια τεράστια οικονομική κρίση αυτή η πανδημία και νομίζω ότι θα είναι χειρότερα από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Και επομένως είναι πάρα πολύ λογικό οι κυβερνήσεις ε, να συμβάλλουν όλες ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την οικονομική ανάκαμψη. Θα είναι δύσκολη, ευάλωτη κατάσταση πρέπει να δούμε τι χρειάζεται το σύστημα υγείας, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε και ότι μπορούμε να διατηρήσουμε ευημερία και θέσεις εργασίας. Αυτή λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε αυτές τις ε, συμφωνίες ε, και τα πακέτα για να αντιμετωπίσουμε τη μετάβαση αυτή. Πρέπει να υπάρξει μετάβαση, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη καινοτομία και ανταγωνιστικότητα και επομένως πρέπει να επικεντρωθούμε πραγματικά στα δύο αυτά στοιχεία στη στρατηγική για την οικονομική ανάκαμψη. Οι ε, δέσμοι μέτρων του ε, Eurogroup ε, σίγουρα θα πρέπει να τα υποστηρίξει. Χρειαζόμαστε λοιπόν τις μεγάλες επιτυχίες σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και περιοχών και περιφερειών. Χρειαζόμαστε τα κονδύλια, χρειαζόμαστε μέτρα εκεί που χρειάζονται περισσότερο και φυσικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και με τον κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φανοβερτφέλτ. ακολουθεί για ένα λεπτό η κυρία Ντάλη λέει. Φυσικά Προφανώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προκάλεσε τον ιό, αλλά ο ανελέητος διωγμό ε, δεν μα επέτρεψε να το αντιμετωπίσουμε και δημιούργησε τεράστιε ζημίε. Αφήνει του εργαζομένου μα ε, χωρί επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό και υποσκάπτει και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνα ε, για τι νόσου και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Όλα αυτά προκάλεσαν ζημία. Για να ανταποκριθούμε λοιπόν σε αυτή την κρίση με προσωρινή αναστολή κάποιων από αυτών των μέτρων, αλλά τελικά να έχουμε και μια από τα ίδια, δεν θα αλλάξει τίποτα. Είναι ε, το αντίθετο της αλληλεγγύης, είναι πραγματικά επιζήμιο και τα 500 εκατομμύρια με πολύ αυστηρούς όρους ε, είναι σαφές ότι ο κάθε ε, πολίτης θα πληρώσει τελικά το λογαριασμό. Ε, αυτό θα είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε ριζικές λύσεις, χρειαζόμαστε αμοιβεποίηση, μηδενικά επιτόκια, πιστοτικές πιστώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σταματήσουμε να συζητάμε ε, για το τι ακριβώ είναι αυτό. Αν πραγματικά χρειαζόμαστε αλληλεγγύη, γιατί δεν έφυγαν οι ετούντε άσυλο από τα ελληνικά νησιά, γιατί δεν μιλήσαμε με τον Ορπάν, γιατί δεν μιλήσαμε κατά των κυρώσεων που είναι ει βάρο των ανθρώπων. Δεν είναι οι Κινέζοι αυτοί οι οποίοι κοσκάβουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι ίδιοι τη συμπολίτε. Ευχαριστούμε κυρία Ντέλη. Ακολουθεί για δύο λεπτά ο κύριο Κάσπαρη. Ακόμη και αν είχαν γίνει τα πράγματα ταχύτερα, εδώ και εβδομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μαλλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένα κράτη-μέλη ε, θεωρούν ότι η Κίνα και η Ρωσία βοηθούν περισσότερο από ότι τα δικά μας κράτη-μέλη. Θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα εκεί που υπάρχει αλληλεγγύα με τους γιατρούς, με τους αναπνευστήρες, με τον προστατευτικό εξοπλισμό και δισεκατομμύρια χρήματα είναι η Ευρώπη και θα πρέπει εμείς να σταματήσουμε αυτή την παραπληροφόρηση ε, να θεωρούμε ότι έρχεται μεγαλύτερη βοήθεια από κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μαχηθούμε να θα δω... Μην θεωρούμε ότι έρχονται χρήματα χωρίς προϋποθέσεις από άλλα κράτη-μέλη. Όταν εντός του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών θεσμών θέλουμε να έχουμε ένα κοινό σχέδιο ανοικοδόμησης της οικονομίας και των κρατών, αυτό θα χρειάζεται μια κοινή διαδικασία όπου κανένας δεν θα παραβλεφθεί, δεν θα έχει ε, προνόμια. Όλοι μαζί θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια κοινή οδό ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά μέτρα ενός κράτους μέλους δεν θα ε, αξιοποιούνται πολιτικά. Και δεύτερον, θα ήθελα να παρέχουμε την απαραίτητη βοήθεια στους πολίτες μας γρήγορα και όσο πιο γρήγορα να επανέλθουμε στις προσωπικές ελευθερίες. Για μένα είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το ψήφισμα που θα ψηφίσουμε η Ευρώπη να μπορεί να λειτουργήσει όλοι, να ε, συνεχίσει να ξανανοίξουν τα σύνορα για την κυκλοφορία των εμπορευμάτων και όταν αύριο θα αποφασίσουμε να υπάρχει κάποια αποθήκευση δεδομένων, αυτό να μην σημαίνει ότι θα μπορούν να μας μπλοκάρουν η Apple, η Microsoft ή να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μας ε, περισσότερο από ότι οι δημοκρατικά ε, εκλεγμένοι μας θεσμοί. Να, μην μπορούν, να μπορούμε εμείς να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα μας καλύτερα από ότι αυτές οι επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Κασπάρη για 1,5 λεπτό ο κύριος Λαρωτηρού. Κυρία Φόντερ Λάιεν, ο Πέτρο Σάνσεθ έχει δίκιο και εσεί έχετε δίκιο όταν λέτε ότι χρειαζόμαστε ένα πραγματικό σχέδιο Μάρσαλ, εάν δεν θέλουμε η Ευρώπη να πέσει σε μια κρίση χειρότερη από το 1929. Το πρώτο σχέδιο Μάρσαλ ήταν 4% του ΑΕΠ των χωρών για πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή καμία χώρα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα μαζικό σχέδιο ανάκαμψη. Καμία χώρα δεν μπορεί να βρει του απαραίτητου πόρου μόνη τη. θα είναι πολύ μικρής διάρκειας και δύναμης αυτά τα σχέδια. Η Ευρώπη λοιπόν είναι η λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να βρεθούν καινούργιοι πόροι. Να θυμηθούμε τι έκανε ο Ρούσβελτ όταν έφτασε στην εξουσία. Η Ευρώπη, η, χώρα μάλλον, οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν σε καταστροφική κατάσταση. Αποφασίζει να τριπλασιάσει τον ομοσπονδιακό προπολογισμό ο Ρούσβελτ τότε. Σε λίγα χρόνια. Θέλει ένα προπολογισμό ισορροπημένο κύριο Ρούσβελτ όμω και ένα ισορροπημένο προπολογισμό δημιουργεί νέου πόρου. Δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό φόρο πάνω στα κέρδη, πάνω στου πιο πλούσιου. Το πρώτο έτο δεν δίνει τίποτα βέβαια ε, και δημιουργεί ε, και δανείζεται με ομόλογα. όμω, επειδή ο φόρο αρχίζει να αποδίδει μετά από 2-3 χρόνια εξισορροπείται ε, ο προπολογισμό. Πρέπει να βρούμε λοιπόν νέου πόρου. Όταν ήμουν μικρό. ήταν 45% ο φόρο στα κέρδη και είναι στο 20% σήμερα. Έχει διαιρεθεί δια δύο ενώ έχουν αυξηθεί τα μερίσματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα φόρο στα κέρδη, ε, ένα, μια μικρή επιβάρυνση πάνω στις, στις χρηματιστηρικές συναλλαγές οι ίδιες χώρες ε, ζητούν να προχωρήσουμε πιο σύντομα στο πράσινο, για το πράσινο deal. Το ίδιο θα, θα πούν ναι, ε, και για ένα σχέδιο Μάρσαλ ε, για την απασχόληση. Να είστε λοιπόν θα λέει κυρία Φοντερ κάντε ό,τι και ο Ρούσβελτ. Ευχαριστούμε κύριε Λαροτερού. Ακολουθεί για δύο λεπτά ο κύριος Φερχόφστατ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στην ε, κυρία Βαντερλάιν, την πρόεδρο της Κομισιόν, αλλά δεν είναι πια εδώ. Γιατί, Γιατί πιστεύω ότι πολύ σωστά αναφέρθηκε στα καθήκοντα που εκπληρώνουν ε, οι γιατροί μας και οι νοσοκόμες μας. Αλλά ε, και εμείς οι πολιτικοί πρέπει να πληρούμε τα καθήκοντα. Το κάνουμε, δεν είμαι βέβαιος. Εδώ και εβδομάδες δεν κάνουμε παρά να συζητάμε για αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ και η ερώτησή μου είναι τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. γιατί δεν το παρουσιάζει αυτό το σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάκαμψης των 3 εκατομμυρίων. Τι περιμένει το Ευρωσυμβούλιο. Θα περιμένει καμιά οκταετία, όπως συνέβη με την Τραπεζική Ένωση, γιατί ακόμη δεν έχουμε Τραπεζική Ένωση. Το Συμβούλιο παίζει πινκ-πονγκ το Φεβρουάριο στο Eurogroup δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για αυτό το σχέδιο και το, στείλα, το στείλατε στο, το για το Συμβούλιο μετά στο Eurogroup το Eurogroup τον Απρίλιο πριν λίγες μέρες πάλι δεν συμφώνησε για ένα κομμάτι του σχεδίου και το ξανά στείλε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μήνυμα μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτό πρέπει να σταματήσει έχετε το δικαίωμα πρωτοβουλίας αναλάβετε τις ευθύνες σας και προτείνεται αυτό που σας ζητά ολόκληρη ολομέλεια εδώ ένα σχέδιο 3 για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση χωρίς ε, καταμερισμό των ε, χρεών με καταμερισμό συγγνώμη των χρεών χωρίς προϋποθέσεις βάσει νέων ιδίων πόρων είναι μια ιστορική εποχή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειαζόμαστε μια πρωτοβουλία τύπου Ντελόρ τον θυμάστε τον Ντελόρ Υπήρχε μια μεγάλη κρίση τότε η οικονομική στασιμότητα και αυτός ξεκίνησε την ενιαία αγορά και μας έβγαλε από την κρίση. Το ίδιο απαιτείται και τώρα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δράσει, όχι να περιμένει να δούμε τα συμπεράσματα ενός Συμβουλίου αναποφάσει του, που δεν θα αποφασίσει τίποτα την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φερχόφσταντ. Ακολουθεί ο κύριος ε, Μπέκ για 3,5 λεπτό. Ε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Προσπαθούμε να βγούμε από μια καταιγίδα. Ε, όταν είχε γίνει Βαστήλη είχαν πει πρόκειται για μια επανάσταση. Και τώρα συζητάμε το Ιανουάριο συζητούσαμε την Πράσινη Συμφωνία να σώσουμε το κλίμα, το μέλλον της Ευρώπης. Το Φεβρουάριο ε, τη ε, ίσα δικαιώματα των φίλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μαδαγασκάρη. Περιμέναν ε, τότε στη Μαδρίτη είχαμε ελάχιστους άρρωστους το Φεβρουάριο άσυλο, η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά είναι συλλογικά συμπτώματα μιας ε, νευρωτισμού, ενός νευρωτισμού. Για αυτές τις φαντασίες ε, παγκυριαρχίας, ε, κυριαρχίας, ενώ η Ευρώπη ολίσθενε μέσα στην αρρώστια η κρίση του κορώνα μας δείχνει ότι η Ευρώπη είναι ασθενής και επιρρεπεί στις ασθένειες. Εδώ πεθαίνουν αναλογικά περισσότεροι άνθρωποι από οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Στην Ιαπωνία, στην Ταϊβάν, στην Νότια Κορέα. Παρότι ήταν εστίες μόλυνσης, πολύ γρήγορα έκλεισαν τα σύνορα, έδωσαν μάσκες, έκαναν τεστ και έτσι πέθαναν λιγότεροι άνθρωποι. Και οι οικονομικές ζημίες είναι πολύ μικρότερες. Ελάχιστου ε, ασθενείς είχε και η Ανατολική Ευρώπη του Ορμπάν και των άλλων, οι οποίοι έκλεισαν τις χώρες τους. Ε, η Δυτική Ευρώπη αντιθέτως ε, απέτυχε. Οι προειδοποίησεις δεν εισακούστηκαν, δεν έκλεισαν τα σύνορα, δεν έδωσαν προστατευτικά ε, ηματισμό και δεν τα έστεραν κανέναν, ούτε τους ε, πρόσφυγε που εργάζονται. Οι πρωθυπουργοί δεν ήξεραν τι να κάνουν, ούτε οι υπουργοί. Ο ένα πήγαινε να ακούσει τον άλλο και έλεγαν όλοι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Γιατί να ακούσουμε αυτούς που λένε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα χρέη. Χρειαζόμαστε την ε, πολιτική ε, αυτή για την υγεία και τους φόρους γιατί για να μπορέσουμε να φτιάξουμε χρέη κοινά για όλους μας. Ο, καθένας έχει τις δικές του ανάγκες ε, και θα πρέπει να δρά ανάλογα. Ε, θα πρέπει να τυπώσει χρήματα η Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική Τράπεζα, λένε αυτά είναι τρέλα. Εναρμονισμός, βελτιστοποίηση, να τα κάνουμε όλα σοσιαλιστικά. Δεν θα φτάνουν αυτά τα χρήματα. Πώς ε, χρεοκοπεί κανείς είχε πει ο Ernest Hemingway πρώτα αργά και μετά ξαφνικά θα αποκαταστήσουμε την υγεία μας όχι ε, με κατάρες προς την ασθένεια αλλά με την καλλιέργεια του δικού μας κήπου ο καθένας και όχι των κοινών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπέκα. Ακολουθεί ο κύριος Έπινγκ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε την όλη συζήτηση για τα ευρωμόλαγα. Το Eurogroup ε, τι κάνει, τσακώνονται σαν τα κοκόρια. Δεν κατηγορώ τους Ιταλούς, τους Γάλλους, τους Ολλανδούς, τους αγαπώ όλους. Αυτοί που φταίνε είναι η Ευρωζώνη, διότι το πρόβλημα της Ευρωζώνης είναι το ίδιο το ευρώ, κύριε Φερχόφσταντ ένα νέο νόμισμα στην ουσία δεν ε, προσφέρει ενότητα. Είναι μια ψευδέστηση. Ξέρετε, φέρνουμε πολλές χώρες μαζί με ένα ενιαίο νόμισμα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στην ιστορία γιατί είναι τεράστιες οι διαφορές και το ευρώ τις κάνει ακόμα μεγαλύτερες και το αποτέλεσμα είναι λογομαχίες παντού, μεταξύ κρατών μελών, εντός κρατών μελών, ε, πικρίες, ακισμοί. Κύριε Φερχόφστετ, ε, μιλάτε με μεγάλο πάθος και ζητάτε ευρωπαϊκό φόρο, αλλά μετά θα ακολουθήσουμε την άγουσα που μόλις μας εξήγησε ο κύριος Μπέκ το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ευρωζώνη δεν νομίζω ότι μπορεί να γεφυρωθεί. Η Ευρωζώνη είναι ε, φυλακή για διάφορους λόγους. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργό είπε ότι οι κάτω χώρες δεν συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης επιφάσεων ε, πλέον. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την πρότασή τους, αλλά ουσιαστικά τι είναι, χρέος, επινέου χρέος, επινέους χρέος. Δημιουργείται ένας χάρτινος ε, ε, πύργος και ένας πύργος της Βαβέλ. Ξέρετε πώς κατέληξε ο πύργος της Βαβέλ. Ο κύριος Γουάλλας, ο COVID-19 πραγματικά ε, έριξε φως στι μεγάλες ανισότητε. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Η πρόεδρο είπε, ε, Βαντερ ότι μόνο αν ε, έχει νόημα η συγγνώμη μας ε, μπορούμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Υπάρχουν οι σημαντικοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας τι θα κάνουμε για όλα αυτά τα χρόνια τους, τα οποία δεν τους πληρώναμε ε, αρκετά. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στα ε, όσα είχαμε προηγουμένως, γιατί ο νεοφιλελευθερισμός ε, θα πριτανεύσει και είναι και η αιτία κάθε κακού για την Ιταλία, για την Ιρλανδία και άλλου. Η Γερμανία και κάτω χώρε έκλεισαν ε, την πόρτα στα μούτρα μα ε, για τον κορονοϊό, αναφέρονται στην αλληλεγγύη, αλλά δεν κάνουν τίποτα για αυτήν. Ε, η Ευρωζώνη λοιπόν μπορεί να υποστηρίξει μόνο τι ισχυρε χώρε. Πρέπει να επιβιώσει, αλλά πρέπει να αλλάξει, πρέπει να πει αντίο στον νεοφιλελευθερισμό. Το ψήφισμα ζητάει να καταπολεμηθεί ο ιό μέσω ε, ε, να σταματήσουμε να υπάρχει και ρωσική ε, και κινέζικη προπαγάνδα. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τους ενήλικου στο δωμάτιο. Ευχαριστούμε κύριε Γουάλλας. Για δύο λεπτά ο κύριος Ντέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε ξανασυναντήσει τέτοια κρίση. Είναι μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Και αυτός ο ιός ε, δεν ξεχνάει κανέναν. Αναγκαστήκαμε να, να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, ε, να επιβραδύνουμε το ρυθμό ζωής μας, ε, να είμαστε μακριά από αγαπημένα μας πρόσωπα, παρότι μας χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Και τώρα χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε την κρίση του κορονοϊού. Όμως από ό,τι φαίνεται ακόμα και σε αυτές τις στιγμές κάποιοι επιτίθενται σε εθνικές κυβερνήσεις ε, ότι είναι, αυτο, ε, ότι είναι ε, αυταρχικές και ότι καταργούν το κοινοβούλιο η Ουγγρική κυβέρνηση και το Ουγγρικό κοινοβούλιο εργάζονται πλήρως Αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου το 90% των Ευρωβουλευτών δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Η, Ευρωπα... η Ουγγρική κυβέρνηση έδρασε όπως το προβλέπει το Ουγγρικό Σύνταγμα για να προστατεύσει τους πολίτες τη και να μπορέσει να αποσυμπιέσει την Ουγγρική οικονομία. Και λάβαμε εντολή από το Κοινοβούλιο για να το κάνουμε αυτό και από το Συνταγματικό Δικαστήριο το οποίο παρακολουθεί την όλη διαδικασία. Αυτά δεν θα πρέπει να είναι τώρα στην ημερήσια διάταξη εδώ. Η κρίση πρέπει να είναι στην ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους τις χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντέλη. Ακολουθεί για ένα μισή λεπτό η κυρία Ρέγναρ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερος ε, μεταξύ άλλων την αδερφή τη κυρία Ντελάγκε βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της πανδημίας και ευχαριστούμε πολύ όλους όσους εργάζονται ακόμα καθημερινά και παρέχουν υπηρεσίες ε, ούτω ώστε να παρέχονται οι βαρισικέ υπηρεσίες. Ε, αυτό δείχνει αυτή η κρίση. 25% 75% ε, είναι γυναίκες αυτές που ε, εργάζονται σε σημαντικές ε, συστημικά θέσεις. Μιλάμε για γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή ε, και τις άλλες που μένουν στα σπίτια τους και αυτές είναι σημαντικές οι γυναίκες δείχνουν ότι είναι ρεαλίστριες λειτουργούν γρήγορα και αμέσως ε, και προστατεύουν και τα παιδιά από την ενδοικογενειακή βία. Πολλές γυναίκες εργάζονται και εκτός ε, και μετά πάνε στο σπίτι και εργάζονται και εκεί. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα ώστε όλα αυτά τα πρακτικά προβλήματα της κοινωνικής αβεβαιότητας να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Η κρίση αυτή λοιπόν είναι θηλυκή, έχει θηλυκό χαρακτήρα, το είπαν τα Ηνωμένα Έθνη. Οι γυναίκες ε, κινδυνεύουν περισσότερο από τον COVID-19. Ε, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα της ενδοικογενειακής βίας. Ε, πρέπει να τα προσέξουμε αυτά μετά από την οικονομική κρίση σώσαμε τράπεζες για να σώσουμε την πραγματική οικονομία, πραγματική οικονομία και τους υπαλλήλου τους. Τα ευρωομόλογα δεν είναι μια αρχή, χρειαζόμαστε και αλληλεγγύη και ενότητα και ένα μεγάλο ιδεώδες. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρέγνερ. Ακολουθούν για δύο λεπτά η κυρία Παγκάζα Ουρτουντούα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούστηκε, ε, ακούστηκαν συγγνώμες. Πολύ καλά. Έγινε αναφορά στους ήρωες, στα θύματα. Έπρεπε να γίνει. Όμως πρέπει να δώσουμε και απαντήσεις. Αυτό είναι υπεραπαραίτητο. Ιδάλλως δεν θα υπάρξει μέλλον για κανέναν. Είμαστε πολύ μικροί, πολύ ευάλωτοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να καταφέρουμε να βγούμε από αυτά ε, μόνοι μπορέσαμε να βγούμε από τα συντρίμια του πολέμου. Οι πρόγονοί μας δημιούργησαν αυτά τα όργανα, αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άνθρωποι, εχθροί, οι οποίοι θα αποφεληθούν την αδυναμία μας. Αν ακούσουμε ε, τις ειρήνες ε, των φανατικών, της, ε, των ταυτοτικών εθνικιστών, θα χαθούμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μηχανισμό που έχουμε στη διάθεσή μα για να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση αλλά και την οικονομική που ακολουθεί. Δεν μπορούμε ε, να μην κάνουμε την κάθε προσπάθεια πρώτα απ' όλα για να σώσουμε ζωέ και μετά για να σώσουμε θέσει απασχόληση, ελευθερίε και ένα σχέδιο για το μέλλον των νέων μα. Η, η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε σε μια σειρά από μέτρα. Η συμφωνία τη Ευρωγκρουπ είναι καλή προς τη κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί για να αντιμετωπίσουμε τις πληγές που έχουν δημιουργηθεί. Χρειαζόμαστε ένα μαζικό σχέδιο οικονομικής ανοικοδόμησης που να χρηματοδοτείται μερικώς από υπάρχοντα μέσα αλλά και μέσω αυτών των ομολόγων ανάκαμψης που θα εγγυάται, θα εγγυάται ευρωπαϊκός προπολογισμός. Πρέπει να γράψουμε ιστορία. Δεν μπορούμε ε, να μην το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να δράσουμε με έναν τρόπο έτσι ώστε η Ευρώπη να εγκαταλείψει αυτό, ε, αυτή την προσέγγιση ε, του τι δανείζουμε ένα στον άλλον. Πρέπει να δράσουμε από κοινού. Οι, οι πρόγονοί μας δημιούργησαν αυτά τα όργανα και πολλοί από αυτούς σήμερα πεθαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουμε πολιτικές για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Να μην χρειαζόμαστε ε, ήρωες, να μην χρειαστεί να κλαίμε θύματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Παγκαζόρτουντούα για ένα λεπτό ο κύριος Γκόκινγκ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ήθελα να τονίσω ότι φυσικά οι σκέψεις μου πάνε στα πολλά θύματα και σε όσους βοηθούν σε κάθε χώρα τους ανθρώπους. Τώρα πάμε σε αυτό που πρέπει να ψηφίσουμε, δυστυχώς. Εγώ θα καταψηφίσω για, πολλούς λόγους όπως είδαμε και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία και στις εκλογές ε, δεν μπορούμε να τιμωρούμε αυτούς που έχουν εκλεγεί. Εδώ χρειαζόμαστε ένα εργαλείο το που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την κρίση του κορώνα. Όχι κάτι άλλο. Τα άλλα είναι πολύ σημαντικά αλλά μπορούμε να τα δούμε αργότερα και να τα συζητήσουμε αργότερα και να τα επεξεργαστούμε αργότερα. Πρέπει να βλέπουμε προ τα μπρο και όχι προ τα πίσω. Πώ θα χρηματοδοτήσουμε τα πράγματα, πώ θα δώσουμε τα μέσα, θα φτιάξουμε του ακρογωνίου λήθου, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τι οικογένειε, ε, να καλύψουν οι οικογένειε ε, τα κόστη για τα παιδιά του, την εγγύηση για τα παιδιά για την οποία μίλησε η Βαντερ Λάιεν. Να βοηθήσουμε την αγοραστική δύναμη, να δώσουμε χρήματα στου ανθρώπου στι οικογένειε τη Ευρώπη ε, που τα χρειάζονται. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση. Σας ευχαριστώ. δυστυχώ ένα λεπτό δεν είναι πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γκόκινγκ. Ε, να πω ότι αυτό το ένα λεπτό δεν το αποφάσισα εγώ, το, η ομάδα σας το ζήτησε. Λοιπόν, για δύο λεπτά η κυρία Περέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, γράφουμε τις σελίδες των βιβλίων της ιστορίας που θα διαβάσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή η Ήπειρος της Ευρώπης ε, φαίνεται να είναι πολύ αδύναμη, ε, ευάλωτη, απειλείται από εθνικισμούς. Και ποια θα είναι ε, το κληροδότημά μας, ε, ενότητα ή διχασμός, ε, γραφειοκρατισμός, γραφειοκρατικός μηχανισμός ή ελπίδα. Θα υπάρχει κάτι καλό για το Βορρά, για τη Βαλτική, για τις χώρες του Νότου. Όχι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιε προκλήσει αυτή τη στιγμή. Ένα ιό ο οποίο διασχίζει σύνορα χωρί ε, κανένα πρόβλημα. Έχουμε τι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε αμφισβητούν τι σχέσει και του δεσμού που έχουμε χτίσει εδώ και δεκαετίε. Έχουμε μια απειλή η οποία ήρθε από την Κίνα, ε, σε οικονομικού όρου όμω. Ε, και επομένω, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε μονιασμένοι σε ένα κόσμο με τόση αβεβαιότητα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη βεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό το καλύτερο που μπορούμε να προσφέρουμε, αυτές οι έρηδες και αυτοί οι διχασμοί. Ο Φράνσις πολύ σωστά είπε ότι πλέουμε όλοι στο ίδιο καράβι και το να ασχολούμαστε μόνο με το δικό μας το μερίδιο δεν θα μπορέσει να σώσει ούτε εμάς αλλά ούτε και κανέναν άλλον από μόνοι μας ως άτομα είμαστε ευάλωτοι και ευπαθείς ως ένα κλαδί ενός δέντρου. Αλλά ενωμένοι θα είμαστε ισχυροί και θα αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Η Ευρώπη είναι το καλύτερο μέρος του κόσμου για να ζει κανεί. Επομένως θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς οι οποίοι χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας. Ε, νέοι, άνεργοι, ηλικιωμένοι, ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για να ε, κρατήσουν ζωντανέ τις επιχειρήσεις τους. Ας δημιουργήσουμε ελπίδα και στην την εξαπλώσουμε. Ας μην επιτρέψουμε στην Ευρώπη να γίνει άλλο ένα θύμα αυτή τη κρίση. Ευχαριστούμε κυρία Περέρα. Τώρα συνάδελφος Σίλβα Περέρα. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μεγάλο άγχος στην ευρωπαϊκή οικονομία. σαν να μας χτύψει ένα, ένα τσουνάμι από όλες τις κατευθύνσεις όμως. Διαπιστώνουμε ότι αυτό είναι απλώς ε, η κορυφή του παγόβουνου. Είναι ε, ένα τεράστιο κύμα το οποίο θα μας χτυπήσει ε, οι θέσεις απασχόλησης, οι επιχειρήσεις, οι οικογένειες. Αν δεν μπορέσουμε να δράσουμε τώρα με αποφασιστικότητα και ισχύ, θα μας χτυπήσει με όλη του τη δύναμη. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτό το κοινό ψήφισμα. Υπάρχει ένα σαφές μήνυμα προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και ένα μήνυμα ε, για τις ε, λίγες αυτές κυβερνήσεις οι οποίες ε, δεν επιτρέπουν να προχωρήσει αυτή η μεγαλύτερη ένδειξη αλληλεγγύης. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας και πρέπει να ε, υπάρχει και κατάλληλη χρηματοδότησή του. Γι' αυτό ακριβώ και χρειαζόμαστε ένα πολιετέ δημοσιονομικό πλήσιο το οποίο δεν θα χαρακτηρίζεται από περικοπέ αλλά από αυξήσει. Και πρέπει να υπάρχει και αυτό το ομόλογο ανάκαμψη. Ομόλογα τα οποία θα εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα ε, υποστηρίζονται και θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτά τα μέσα και τα μέτρα. Δεν μπορούμε απλώ ε, να ε, μπούμε χωρί κανένα μέτρο στην επόμενη κρίση. Χρειαζόμαστε να ακούσουμε και τη μας λένε οι πολίτες ότι δεν θα δεχτούν πλέον ε, εθνικούς εγωισμούς οι οποίοι θα είναι εις βάρος ε, της Ευρώπης. Εγώ είμαι με το λαό και θέλω να εργαστώ για αυτόν. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Σίλβα Περέρα για δύο λεπτά. Ακολουθεί ο συνάδελφος κύριος Κνότεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω το σεβασμό μου προς όλους όσους συνεισφέρουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση. Στο πρώτο μέρος της συνεισφοράς μου θα ήθελα να υποστηρίξω το πακέτο που παρουσιάζει η Κομισιόν για την μετωπίση του κορονοϊού. Προετοιμάστηκε γρήγορα και σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Ρέτζη του Κοινοβουλίου και αναφέρεται σε μέτρα ε, τα οποία αντιμετωπίζουν τις ανάγκες ε, των συμπολιτών μας. Ευχαριστούμε για αυτή τη συνεργασία. Στο δεύτερο μέρος θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σας σε δύο σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται με βάση το COVID μέρος στο τομέα τη ενέργειας και της βιομηχανίας αυτή τη στιγμή έχουν ζήτημα επιβίωσης. Θέλουμε να μειώσουμε ε, τις, εκπομπές δεξιού του άνθρακα ε, και ταυτόχρονα να έχουμε ε, το COVID αυτό είναι ένα μείγμα το οποίο είναι καταστροφικό, εκρηκτικό. Φανταστείτε βιομηχανικές περιοχές που είναι και τουριστικές. Θα πρέπει να ανακάμψουν οι βιομηχανίες μας ε, για να μπορέσουμε στη συνέχεια ε, να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική ε, μετάβαση. Σας ζητώ λοιπόν βραχυπρόθεσμη κατάργηση του συστήματος ενταλλαγής εκπομπών για δύο χρόνια έτσι ώστε να μην χαθούν θέσεις απασχόλησης, να μην χαθεί ενέργεια, να σταθεροποιήσουμε περιφέρειες και βιομηχανίες, ε, να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση και έτσι να σέβονται γι' αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, και στο ευρωπαϊκά ΣΠΑ που συνδυάζουν την υγεία και τον τουρισμό. Μπορούν να βελτιώσουν αυτά τη δημόσια υγεία και μετά την επιδημία του COVID. Ο τομέας ΣΠΑ αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τεράστιε δυσκολίε και χρήζει υποστήριξη. Στην πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η πρωτοβουλία τη Επιτροπή προ την κατεύθυνση αυτή θα ήταν εξαιρετικά καλοδεχούμενη. Ευχαριστούμε κύριε Κνότεκ. Ακολουθεί για ένα λεπτό ο κύριο Φιντάντσα. Ευχαριστώ πρόεδρε από αυτή την κρίση δεν πρόκειται να βγούμε με κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας ωραίες προτάσεις ε, και φάση 2. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες και να ανταποκριθούμε άμεσα αυτό που δεν έγινε στην αρχή όταν θεωρούσαμε ότι ο COVID-19 ήταν απλά ένα πρόβλημα της Ιταλίας. Τώρα ε, χρειαζόμαστε ευελιξία για τους δημοσίου λογαριασμούς, τις ε, κρατικές ενισχύσεις ε, και τα διαρθρωτικά ταμεία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιτέλους κάνει τη δουλειά της μετά από την ντροπιαστική της συμπεριφορά. Τώρα για το επόμενο συμβούλιο, το πακέτο που υπάρχει πρέπει να πούμε σαφές. το Ταμείο Ανοικοδόμησης, ναι, και τα αλλά όχι στο μέσο οικονομικής σταθερότητας. Θα πρέπει να βγούμε από την κρίση για το πράσινο η συμφωνία. Δεν θέλουμε άλλα κόστη για τις ε, επιχειρήσεις μας που υποφέρουν από την κρίση. Ναι, μόνο σε ενάρετες επενδύσεις και τέλος να υπερασπιστούμε τα σύνορα, διότι ενώ κλείνουμε τους Ευρωπαίους στα σπίτια τους δεν γίνεται να συνεχίζουν να λιμένονται όλοι στην ε, Μεσόγειο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Φιντάντσα για δύο λεπτά. Ο συνάδελφος κύριος Πέτερς. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καθημερινά πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι στα νοσοκομεία μας, στις οίκους ευγυρίας ή στο σπίτι τους. Δεν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, πώ γίνεται κάποιε χώρε χώρες να μην δείχνουν αλληλεγγύη και πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Αυτό το κοινοβούλιο σήμερα και αύριο θα δείξει στους Ευρωπαίου σαφώ ότι από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι υπάρχει αυτό το κοινό ψήφισμα με όσο γίνεται ευρύτερη πλειοψηφία και να ψηφιστεί με όσο γίνεται ευρύτερη πλειοψηφία. Υποστηρίζουμε λοιπόν αυτό το ψήφισμα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση ενωμένη. Να δράσουμε στον τομέα των συστημάτων υγείας, να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους, τους εργοδότες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να είμαστε αποφασιστικοί. Χρειαζόμαστε τα ευρωομόλογα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και να πούμε ότι κανείς δεν φταίει για αυτή την κρίση και βεβαίως συνεργαστούμε περαιτέρω για το Green Deal αλλά και για μια, μια νέα βιομηχανική ε, πολιτική ε, την κυκλική οικονομία, βιώσιμη γεωργία ελπίζω μετά από αυτή τη συζήτηση αλλά και τη συζήτηση των τροπολογιών θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει να τα εφαρμόσουν από εκεί πέρα όμως προς όφελος όλων μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Πέτερς. Ακολουθεί για ένα μισή λεπτό η κυρία Σπούρεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μπορούμε καρδερκα μια πανδημίας που θα, θα ακολουθήσει μια οικονομική κρίση, όπου πεθαίνουν άνθρωποι, όπου χάνουν τις θέσεις εργασίας τους, ε, όταν το οικονομικό προσωπικό ε, δίνει μάχη καθημερινή με την πανδημία με λίγα μέσα δεν μπορούν κάποιες χώρες να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία αυτή ε, για να φημώνουν τη δημοκρατία. Όταν ο Βίκτορ Ορμπάν στην Ουγγαρία περιορίζει τα δικαιώματα ε, των LGDPI, LGBTI, των ΛΟΑΤΚΙ, αλλά και στην Πολωνία πρέπει να αντιδράσουμε. Ήδη στην Πολωνία ε, είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση στην ε, άμβλωση σε ε, μέσα περιορισμού των γεννήσεων αντισυλληπτικά θα πρέπει λοιπόν να είναι μια προτεραιότητα και αυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Είναι η βάση των αξιών μας το να περιορίζουμε το δικαίωμα στην άμβλωση. Ήδη επηρεάζει τις γυναίκες που ήδη υφίστανται διακρίσεις, που ζουν στην εξοχή, στην ε, επαρχία, που δεν έχουν μέσα, που δεν είναι ανεξάρτητες. Εάν δεν το επιλύσουμε το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων με διαφορετικά δικαιώματα για τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Πρέπει όλοι να έχουμε τα ίδια δικαιώματα όπου και να ζούμε. Ευχαριστούμε κυρία και για δύο λεπτά. Ο κύριος Πισλάρου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε πολύ για αλληλεγγύη. Δυστυχώς η αρχή της αλληλεγγύης θα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη. Δεν είναι απλά ρητορία. Πρέπει πραγματικά να βοηθήσουμε ένα τον άλλον. Υπάρχουν, υπάρχουν δείγματα αλληλεγγύη στι κοινότητε μας. Χρειάζεται αλληλεγγύη μεταξύ διαφόρων περιφερειών τη ίδια χώρα, αλλά και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η προσπάθεια αλληλεγγύη αποτελεί μέρος της ουσίας της Ένωσης. Είναι οι αξίες που ορίζουν την Ένωση. Η κρίση βεβαίως μας επηρεάζει όλους. Δεν έχουμε όμως όλοι τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια μέσα για να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις που προκύπτουν. Διότι 22% του πληθυσμού της Ένωσης κινδυνεύει με κοινωνικό αποκλεισμό και με φτώχεια. Και 25% των παιδιών που ζουν στην Ένωση. Αυτή η κρίση μπορεί να επηρεάσει πολίτες ανά την Ευρώπη, αλλά επηρεάζει συχνά και πλήττει ανθρώπους που είναι αόρατοι στην κοινωνία μας. Σε, μια σε, σε σπίτια όπου υπάρχει υπερπληθυσμός δεν μπορεί να υπάρξει ε, κοινωνική απόσταση δεν υπάρχουν διακρίσεις ό,τι αφορά την πρόσβαση στην πληροφορία, σε βασικές υπηρεσίες. Οδηγούν τους ανθρώπους αυτές οι διακρίσεις σε περαιτέρω αποκλεισμό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, ε, πανδημία. Εμείς θα ψηφίσουμε ε, το, την τροπολογία του 2023 για να δοθούν χρήματα από το ανάλογο ταμείο προς τους πιο αδύναμους. Ε, θα χρειαστούν θα χρειαστεί περαιτέρω χρηματοδότηση με θα πρέπει να σταματήσει η γραφειοκρατία, να αλλάξουν οι κανόνες χρηματοδότησης. Αυτό θα πρέπει να τα πούμε μετά στου Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πεσλαρού. Ακολουθεί για ένα λεπτό κύριο Ρόος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κρίση του κορονοϊού οδήγησε σε πάρα πολλά θέματα και απειλεί να ε, καταστρέψει την ευρωπαϊκή οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου των Νόσων, το ECDC, είναι μια υπηρεσία που στόχο έχει να αυξήσει την ευρωπαϊκή άμυνα ε, σε ε, μεταδοτικές νόσους. Το ECDC στις 12 Ιανουαρίου έδωσε προειδοποίηση και είπε ότι είναι μεγάλη η πιθανότητα να υπάρξει ε, πανδημία και περαιτέρω εξάπλυση του κορονοϊού και η εμφάνιση του ιού σε ένα κράτος μέλος χωρίς προληπτικά μέτρα θα έχει τεράστιες συνέπειες, ολέθριες συνέπειες. Το ECDC λοιπόν σε διάφορα επίπεδα, σε καθημερινή βάση ήρθαν σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ στραβά σε θέματα πρόληψης. Δεν υπήρχε άμεσο κλείσιμο των συνόρων σε, από περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, δεν υπήρχε εντοπισμός ε, ασθενών που έρχονται από αυτές τις περιοχές, ε, επιβατών μάλλον που έρχονται από αυτέ τι περιοχέ και φυσικά οι συνέπειε ήταν ολέθριε. Θα ήθελα να ζητήσω από τη Στέλλα Κυριακίδη, λοιπόν, που είναι υπεύθυνη για τα θέματα αυτά, να αναλάβει τι ευθύνε τη, αν όχι να παραιτηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρώσο. Ακολουθεί για δύο λεπτά ο κύριος Χάνσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το COVID-19 είναι καταστροφή σε ανθρώπινη, κοινωνική και ε, οικονομική κλίμακα και πλήττει φυσικά πορούς από μας. Πέρα από τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από τον ίδιο τον ιό, προβλέπεται και μεγαλύτερη οικονομική κρίση από την 1929 ε, ε, ε, και το κράχ. Επομένως, περιμένουμε ύφεση της τάξης 13 και 32% ο ΙΕΔ κρούει τον να του κινδύνου για επισητιστική κρίση. Θα πρέπει επίσης να δούμε και τι γίνεται με το εμπόριο, διότι απειλείται να καταστραφεί η διεθνής αλυσίδα αξιών. Επομένως, όλα αυτά θα είναι και απαραίτητα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα βραχυπρόθεσμα για να μπορέσουμε να έχουμε και φαρμακευτική ε, περίθαλψη για αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερα και για όχι για αυτούς που τα προσφέρουν τα περισσότερα. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά μέτρα, ε, μέτρα μάλλον προστατευτισμού για να προστατεύσουμε αυτούς οι οποίοι ε, πλήττονται από τον ιό. Το εμπόριο σίγουρα είναι τμήμα της οικονομικής ανάκαμψης, επομένως θα πρέπει να τα βάλουμε στο προσκήνιο γιατί αλλιώς θα στερήσουμε ζητήσουμε από πολύ σημαντικές χώρες ε, ένα τομέα ο οποίος το χρειάζονται περισσότερο αυτή τη στιγμή. Στο παγκόσμιο εμπόριο θα πρέπει να έχει στρατηγικά αποθέματα και θα πρέπει να φροντίσουμε να προστατεύσουμε τις αλυσίδες διανομής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να υπερασπιστεί ε, πολυμερείς λύσεις, θα πρέπει να ε, ενισχυθούν ε, οι συμφωνίες του ΠΟΕ για την κατάργηση των δασμών σε φαρμακευτικά προϊόντα και να περιλάβουμε περισσότερα προϊόντα στους καταλόγους. Ε, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πατάξουμε και να κερδίσουμε αυτό τον ιό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χάνσεν. Για ένα μισή λεπτό η κυρία Αρένα. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι καταστρεπτική αυτή η πανδημία για τα μέσα θύματα του ιού, αλλά θα είναι το ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τους Ευρωπαίους πολίτες και πιο ειδικότερα για τους πιο ευάλωτους. Η κυρία Βαντερλάιν το είπε. Πράγματι έχει γίνει ήδη σημαντική προσπάθεια από την Ευρώπη, χάρη στη δική της πρωτοβουλία, αλλά και χάρη στη δική μας υποστήριξη. Είπε όμως επίσης ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και εγώ θα προσέθετα ότι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα και αλλιώ, Όχι μόνο περισσότερα, αλλά και με πιο φιλόδοξο προπολογισμό, περισσότερα και με καταμερισμό του χρέους που είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε τον οικονομικό και κοινωνικό κλειδονισμό. Αλλά όπως είπαν όλοι, η λέξη κλειδί είναι η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι το αντίθετο της λιτότητας, θεωρώ εγώ. Ξέρουμε όλοι ότι το καλύτερο εργαλείο της ε, αλληλεγγύης είναι το δικό μας σύστημα κοινωνικής ε, ασφάλισης, οι δημόσιες υπηρεσίες μας, αλλά και οι κοινωνικές διαβουλεύσεις ε, για την προσαρμογή των μισθών και την ανακατανομή. Όλα αυτά τα κατέστρεψε η λιτότητα τα τελευταία χρόνια, οπότε πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη θα εκφραστεί επίσης και με μέσω μιας ευρωπαϊκής φορολογίας, φορολογίας πιο δίκαιης, Πρέπει να δώσουμε τέλος σε αυτό το φορολογικό ανταγωνισμό που άδειασε τα εθνικά ταμεία και τα ευρωπαϊκά ταμεία. Επίσης θα πρέπει να υλοποιήσουμε μια αλληλεγγύη εξωευρωπαϊκή διότι παρότι η πανδημία είναι καταστρεπτική για τους πολίτες μας το ίδιο είναι και για τις άλλες υπήρους και θα είναι δραματική η κατάσταση οι συνέπειες για την Αφρική ε, για να υποστηρίξουμε μια ιδέα ακύρωση του χρέου και βοήθειας προς την Αφρική θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε και εκεί τη φοροδιαφυγή και αυτό είναι καθήκον μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Αρενά. Για δύο λεπτά ακολουθεί η κυρία Μέτσολα. Ευχαριστώ. Αυτός ο ιό δεν γνωρίζει σύνορα. Γνωρίζει όμω ήρωε, οι γιατροί, οι νοσοκόμε οι φαρμακοί οι, φα, οι φαρμακοποιοί, οι μεταφορείς, οι ταμείες, τα σούπερ μάρκετ έχουν παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στι δύσκολες συνθήκες και αυτά που είπε ο πρόεδρος Μάιερ είναι πολύ σωστό. Εδώ, αυτό δεν είναι πόλεμος. Εδώ δοκιμάζεται το πνεύμα μας, δοκιμάζεται η ανθρωπιά μας. Δεν πρέπει οι δυναμίες της Ευρώπης ε, να γίνουν πιο ε, εμφανείς με αυτή την κρίση. Πρέπει η, η δύναμη μας να γίνει πιο εμφανής. Έχουν μεταφερθεί ασθενεί από τον Πέργαμο στη Βαβαρία. Ρουμανοί, Ρουμάνοι γιατροί πήγαν στην Ισπανία. Μεγάλοι designers αυτή τη στιγμή ράβουν μάσκες. Θα πρέπει λοιπόν αυτά ε, να τα επεκτείνουμε και σε μια κοινή προσπάθεια και σε μια κοινή προμήθεια για τα εμβόλια όταν θα τα έχουμε. Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή μένουν πίσω και δεν βρίσκουν ε, πού να απευθυνθούν. Πρέπει να φανούμε ευέλικτοι και να συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε για να καλύψουμε και αυτού. Ε, και σε σχέση με την πανδημία του COVID-19 υπάρχει βεβαίω και μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στη Μεσόγειο. Βλέπουμε αυξημένου αριθμού πλοίων που φεύγουν από τη Λιβύη και μένουν στη θάλασσα, δεν μπορούν να αποβιβαστούν. Χρειάζεται μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση. Χρειάζεται μια πραγματική αλληλεγγύη. Πρέπει να σωθούν ζωέ και δεν μπορούμε να αφήνουμε τι χώρε που είναι στην πρώτη γραμμή, όπω η Ιταλία, η Μάλτα, η Ελλάδα, μόνε του. Πρόκειται για μια κρίση όπου η Ευρώπη πρέπει να δείξει την πραγματική φύση τη. Και δεν μπορούμε εδώ να υπολοιπούμεθα, διότι μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Ευχαριστούμε κυρία Μέτσολα για ένα μισή λεπτό κύριο Präsident. Πριν από ένα χρόνο είπα ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι, οι, οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη, διότι αντιμετωπίζουμε κοινέ προκλήσει. Και αυτέ τι προκλήσει μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε ε, μόνο από κοινού. Ενωμένα. Και τώρα έγινε αυτή η τραγωδία ε, Χρειαζόμαστε την τραγωδία αυτή τη δραματικότητα για να καταλάβουμε ότι η κρίση δεν σταματάει στα σύνορα. Πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κρίση από κοινού. Βλέπουμε ποιοι είναι οι τομεί όπου πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε του Ευρωπαίου πολίτε. Επίση, βλέπουμε σαφώ ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επιδείξουν αλληλεγγύη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κινητοποιήσει πόρους ε, για να μπορέσει να απαλύνει τη ζημιά που έχει δημιουργηθεί στον τομέα της υγείας αλλά και στην οικονομία γενικότερα. Δυστυχώς βλέπουμε και κάποια κράτη-μέλη που καταχρώνται της εξουσίας τους και παίρνουν επίγοντα μέτρα όπως στην Ουγγαρία. Ξέρετε τι έκανε στην Ουγγαρία ο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος πλέον μπορεί να πάρει οποιαδήποτε απόφαση ακόμα και αποφάσεις που δεν έχουν καμία σχέση ε, με τον κορονοϊό και την κρίση του κορονοϊού. Δεν δέχεται διεθνείς λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης και βεβαίως πολλοί εργαζόμενοι που έχασαν τη δουλειά τους μένουν χωρίς καμία απολύτως ενίσχυση και βοήθεια από τον κύριο Όρμπαν. Θα πρέπει να προστατευτούν οι πολίτες από τις φυσικές καταστροφές ε, και άλλες ζημιές όμως και θα πρέπει ε, να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστούμε κύριε Ρονά. Για δύο λεπτά η κυρία Βάης. Ευχαριστώ. Όταν ένα επιθετικό ιό επιτίθεται στου πνευμονέ μα και δεν έχουμε καρδιά αρκετά δυνατή, τότε πεθαίνουμε. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί θα χάσει του γονεί του. Και κάποιο άλλο μπορεί να χάσει κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, ένα σύντροφο. Αυτό μα μαθαίνει η COVID-19, αλλά μα μαθαίνει και πολλά περισσότερα. Μιλάμε για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ω πυρήνα τη οικονομία μα και των οικονομικών μας ε, χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων αλλά οι επιχειρήσεις δεν είναι το επίκεντρο μόνο είναι οι πνεύμονες όταν μιλάμε για το κλίμα το... και εκεί αναφερόμαστε σε πνεύμονες μιλάμε για το τι πνεύμονες θα αφήσουμε στην επόμενη γενιά οι πνεύμονες λοιπόν το κλίμα οι πνεύμονες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρειάζονται μια ισχυρή καρδιά για να συνεχίσουν να λειτουργούν ε, ώστε εκατομμύρια οικογένειες να έχουν να φάνε η οικονομία μας και το κλίμα είναι οι καρδιές θα πρέπει να διατηρούν με την ε, επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών. Θα πρέπει οι έρευνες και οι προσπάθειες να γίνουν για να δημιουργήσουμε τον προστατευτικό εξοπλισμό και να τον έχουμε διαθέσιμο. Πρέπει να αυξήσουμε την πράσινη προσπάθεια ούτως ώστε να επιτύχουμε την ουδετερότητα, την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Η καρδιά, λοιπόν, ο πυρήνα για τον οποίο μίλησα, είναι η ενιαία αγορά. Δημιουργήσαμε την ενιαία αγορά για να μην πολεμάμε μεταξύ μας. Η εσωτερική αγορά λοιπόν καθορίζει εδώ τα πάντα μέσω αυτής προστατεύουμε την καρδιά μας η οποία θα πρέπει να χτυπά κανονικά σε αυτή την κρίση χωρίς κανένα εμπόδιο και ουδέτερα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι κλιματικές λύσεις και πρωτοβουλίες που χρειαζόμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο θα έχουν αποτελέσματα για όλο τον κόσμο ούτως ώστε να μάθουμε από την κρίση Ελπίζω ότι μέσω αυτής της κρίσης του COVID θα προστατεύσουμε τη μόνη μας καρδιά, δηλαδή την εσωτερική αγορά. Ευχαριστούμε κυρία Βάης. Ακολουθεί η κυρία Πιτσέρνο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τίποτα, τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Αυτή είναι ε, μια διαπίστωση την οποία κάνουμε όλοι μας, ο καθένας από μας. Τίποτα δεν θα είναι όπως πριν και ισχύει για όλους, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Και επομένως εδώ και τώρα ήγηκε και η ώρα να αναρωτηθούμε μήπως και για την Ευρώπη, ακόμα και για αυτό το μεγάλο όνειρο το οποίο γεννήθηκε από τα ερήπια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πελέμου θα είναι τα πράγματα τα ίδια. Σήμερα συζητούμε για αλληλεγγύη, συνάδελφα θα είναι η αλληλεγγύη, η ένδειξη της Νέας Ευρώπης. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή θα είναι η μεγάλη καινοτομία. Αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την αλληλεγγύη του πιο ισχυρού προς τον πιο αδύναμο. Δεν μπορούμε να μιλούμε για κάτι τέτοιο στο εγγύς μέλλον κανένας ε, δεν θα είναι αρκετά ισχυρός ώστε να μπορέσει να τα καταφέρει μόνος του. Αναφερόμαστε λοιπόν σε μια αλληλεγγύη η οποία θα πρέπει να περιλάβει τους πάντες. Όλα τα θεσμικά όργανα, όλα τα κράτη-μέλη για να υπερβούμε μια κρίση η οποία ελοχεύει ο κίνδυνος ε, να καταστρέψει όλες μας τις οικονομίες, όλες μας τις ελευθερίες ε, και όλα μας τα κοινωνικά δικαιώματα. Περί αυτού πρόκειται. Και επομένως είναι απαραίτητο να επιδείξουμε σθένος, να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο, κάθε νέο μέσο ανύπαρκτο μέχρι τώρα και να το οποίο μας ε, ε, προτείνονται ακριβώς λόγω της αίσθηση του κατεπήγοντος και του θάρρους. Αν λοιπόν ε, δεν μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον αυτό, πραγματικά κύριε Πρόεδρε, τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε κύριε Πιτσέρνο. Ακολουθεί για 1,5 λεπτό ο κύριος Φάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί που είχαν ήδη πολλά. Γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που είπε η συνάδελφος Πιτσέρνο μόλις τώρα Τίποτα δεν θα είναι πια όπως παλιότερα κύριε Πρόεδρε. Αυτό ισχύει για αυτή την κρίση κορώνα. Και έτσι οι συζητήσεις στα κράτη-μέλη και εδώ πρέπει να αλλάξουν. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε λύσεις και όχι μόνο σε παλιότερα προβλήματα που απομένουν ακόμα. Γι' αυτό είναι σωστό αυτό που λέει σήμερα το ψήφισμα που επικεντρώνεται σε δύο σημεία. Πρώτον, στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και δεύτερον, στο ζήτημα του πώς θα βγούμε κοινά μαζί από την κρίση. Θα ήθελα να δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι ότι η κυρία Φοντερ Λάιαν είπε στην αρχή είναι πολύ σημαντικό να αποκαταστήσουμε την εσωτερική ε, αγορά. Αλλά αυτό δεν θα γίνει με όλα αυτά που κάνει η Κομισιόν τι τελευταίε εβδομάδε και λέει τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να έχουν περισσότερη ευελιξία. Και κάθε φορά που εμφανίζεται ένα πρόβλημα στην οικονομία, ρίχνουμε την ευθύνη στα κράτη-μέλη η Κομισιόν δεν μπορεί να λέει ότι όλα είναι καθήκοντα των κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να βρίσκει μια λύση έτσι που τελικά δεν βοηθά κανέναν, δεν βοηθά τον καταναλωτή. Ε, όταν ας πούμε ε, ισχύουν άλλα στη διπλανή χώρα. Οπότε η Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για να τηρηθεί λοιπόν αυτή η εσωτερική αγορά. Το ίδιο ισχύει και για τα φάρμακα. Χρειαζόμαστε μια κοινή έξοδο από την κρίση. Να ανοίξουμε μαζί τις χώρες και μαζί να κάνουμε τον καταμερισμό δεδομένων που, και την κοινή χρήση δεδομένων στην οποία αναφερθήκαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σβάμπ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Γιόντσεβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να έχουμε μια συντονισμένη απάντηση στην πανδημία. Αλλά η κρίση απαιτεί να κάνουμε πολύ περισσότερα και πολύ περαιτέρω. Χρειαζόμαστε ε, συγκεκριμένη ευρωπαϊκή ηγεσία, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανοικοδόμηση της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο ερωτήσεις. Ε, το Σέγγεν, το κράτος δικαίου και την ελευθερία έκφρασης. Στα σύνορα είδαμε και πάλι πάλι ότι η προστασία των συνόρων έγινε μεγαλύτερη από την προστασία της Ευρώπης των Ευρωπαίων πολιτών και των δικαιωμάτων τους. Κλείνουμε ε, τα σύνορα χωρίς μια συντονισμένη προ, ε, στρατηγική και αυτό δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Το κράτος δικαίου. Η κρίση αυτή δεν θα πρέπει να στερεήσει τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να επιλέγουν ε, υγειονομική περίθαλψη ή ανθρώπινα δικαιώματα και η έκκλησή μου δεν απευθύνεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο Συμβούλιο. Ε, θα πρέπει να σπάσει η σιωπή στο Συμβούλιο για το κράτο δικαίου, να κατανομάσουμε το πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε από κοινού. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να ε, πατάξουν και την ελευθερία έκφραση. Σε κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, διώκονται άνθρωποι γιατί εκφράζουν δημοσίω την άποψή του, όπω για παράδειγμα στη Βουλγαρία και όχι μόνον. Ε, Κυρίε και κύριοι, η Ευρώπη πρέπει να δρώσει τώρα. Ω κράτη-μέλη πρέπει να επιβιώσουμε από αυτή την κρίση από κοινού για να μπορέσουμε να σώσουμε την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γιόντσεβα. Ακολουθεί για ένα μισή λεπτό η κυρία Σπυράκη. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε Σεύκοβιτ, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή την κρίση υπάρχουν δύο θέματα τα οποία μπορούν να αναδειχτούν ιστορικοί καταλήτες το πρώτο είναι ο τρόπος που η ευρώπη αντιμετωπίζει τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης. το σχέδιο marshall στο οποίο αναφέρθηκε και σήμερα η κυρία φοντερ λάιεν η πρόεδρος φοντερ λάιεν πρέπει να πάρει αμέσως σάρκα και οστά. άρα για αλήθεια τι περιμένει η κομισιόν για να προχωρήσει και να πιέσει τα κράτη μέλη να πάρουν την απόφαση το ομόλογο της ανάκαμψης που σήμερα ψηφίζουμε και προτείνουμε είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που θα δώσει στις οικονομίες μας τη δυνατότητα για περισσότερη ρευστότητα. μόνο υπερβαίνοντας φόβους και στερεότυπα μόνο ενδυναμώνοντας την παρουσία της ευρωπαϊκής ένωσης μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους πολίτες σε αυτή την πιο σκοτεινή ώρα. και σε αυτή την πιο σκοτεινή ώρα χώρες όπως η πατρίδα μου η ελλάδα έδειξαν πως τα κατάφεραν με πειθαρχία και ισχυρή κυβερνητική καθοδήγηση από τον πρωθυπουργό κυριάκο μητσοτάκη. τώρα όμως χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή στήριξη την ευρωπαϊκή στήριξη που δεν θα θυμίζει μνημόνιο που δεν θα παραπέμπει σε τρόικα και που θα δείχνει αληθινή αλληλεγγύη. η δεύτερη πρόκληση είναι το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που μπορούμε να προχωρήσουμε μετά την κρίση αυτό που θα βασίζεται στον οδικό χάρτη του green deal που θα προβλέπει βιώσιμη ανάπτυξη που θα δίνει έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην κυκλική οικονομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. κυρίε και κύριοι συνάδελφοι το βλέμμα των πολιτών της ευρώπης είναι στραμμένο εδώ. σήμερα οι ορθόδοξοι βιώνουμε το γολγοθά την ημέρα των παθών. είναι χρέος μας να οδηγήσουμε τις κοινωνίες μας τις οικονομίες μας στην ανάταξη που χρειάζονται λαμβάνοντας τα μαθήματα από αυτή την παγκόσμια κρίση σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Σπυράκη. Ακολουθεί για ένα μισή λεπτό ο συνάδελφος κύριος Λόπες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζούμε μια κοινωνική κρίση χωρίς προηγούμενο για αυτή τη γενιά που θα έχει επιπτώσεις καταστροφικές και οικονομικές και κοινωνικές που μας έχει ρίξει στα σκηνιά αλλά μας έχει φέρει μπροστά στον καθρέφτη μας και, και πολλοί Ευρωπαίοι δεν μας άρεσε καθόλου αυτό που είδαμε στον καθρέφτη. Μετά από συζητήσεις, ε, κάποιες πρώτες συζητήσεις που ήταν αρκετά ντροπιαστικέ, το κύριο Γκρουπ έφτασε να κάνει το πρώτο βήμα. Τώρα το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ζητεί ένα πλήρες πακέτο, ένα φιλόδοξο πακέτο στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συνέλθει την επόμενη εβδομάδα. Με ένα μήνυμα σαφές, καθαρό. Δεν παίζουμε μόνο το μέλλον μας ως Ευρώπη. Παίζουμε και την επιβίωσή μας στην διαχείριση αυτή τη κρίση. Η επιβίωση και το μέλλον τη Ευρώπη εξαρτάται από τη δυνατότητα που θα έχουμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό σχέδιο ανάκαμψη για την οικονομία, για αυτήν την Ήπειρο. Ένα σχέδιο ανάκαμψη το οποίο θα σημαίνει ότι θα έχουμε ένα κοινό χρέο, διότι είναι κοινό και το μέλλον μα. Πράσινο σχέδιο ανάκαμψη. Βιώσιμο, για μια βιώσιμη οικονομία Πάντα βεβαίω ο, ο, ο μεγαλύτερο εχθρό μα είμαστε εμεί οι ίδιοι. Ο εχθρό του εαυτού μα είμαστε εμεί. Οι εθνικοί εγωισμοί